Meine sehr geehrten Damen und Herren. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Μογγολίας αγαπητέ Έλμπερκτος. Μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα που μπορούμε να σας καλωσορίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, η Μογγολία η πατρίδα σας είναι ένα κράτος, μια χώρα με παλαιά και πλούσια πολιτιστική παράδοση, με ένα πληθυσμό, με μια δημοκρατία πολύ νεαρή και πολύ ζωντανή, παλόμενη δημοκρατία. Έγιναν το 1989 οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές. Πέρυσι εσείς ηγηθήκατε της ε, διαμόρφωσης μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και μπορέσατε μέσα από μια δύσκολη κατάσταση να βοηθήσετε να βγει η χώρα σας, να έχει μια ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στεναρή η γεωγραφική θέση της χώρας σας μεταξύ των δύο μεγάλων και ισχυρών κρατών, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, είναι ασφαλώς δύσκολη μερικές φορές, το συζητήσαμε και στις δημιουργίες μας συνομιλίες, αλλά καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακά τα επιτεύγματα της Πολωνίας. Γιατί έτσι βλέπουμε πόσο ουσιαστική πολιτική μπορείτε να κάνετε και είναι φάρος στην περιοχή της η Μογγολία κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερω που μπορούμε να υποδεχθούμε σήμερα τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος ε, θα είναι ο επόμενος οικοδεσπότη της Συνόδου Κορυφής Άζεμ το 2016. Πρόκειται για μια σύνοδο πολύ σημαντική για την γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Μια συνόδο στην οποία περιφερειακά και διαπεριφερειακά προβλήματα μπορούν να βρουν λύσεις. Είμαι βέβαιος ότι μπορούν οι συνομιλίες που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα της χώρας σας να οδηγήσουν ουσιαστικές λύσεις. Και εμείς προσβλέπουμε και στην Συμφωνία Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μογγολίας που περιμένουμε να κυρωθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιότιμε κύριε Έλβεν Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξοχότητες κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι απλό.